Αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην χάνουμε χρόνο, γιατί έχουμε διάφορε υποχρεώσεις όλοι μας. Οπότε ας περάσουμε στο πρώτο σημείο, στην ημερήσια διάταξη, που είναι το σημείο αριθμός 31. Θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ευλίν Γκέπαρτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το νέο πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την πραγματοποίηση της ε, ψηφιακής μετάβασης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, της ε, συνολικής ευρωπαϊκής οικονομίας και τη διοίκησης. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια οικονομική και δημοσιονομική βάση η οποία θα στηρίζει πολλές, ε, πολλά σημαντικά έργα υποδομής στην Ευρώπη. Οι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν τη κυβερνοασφάλεια, απόκτηση ενισχυμένων και προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και προηγμένων ε, λύσεων κοινού συμφέροντος. Συνολικά κατατέθηκαν 132 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Οι τροπολογίες αυτές αντικατοπτρίζουν έντανα την ε, θετική στάση της Επιτροπής ε, την ψηφιακή Ευρώπη. Στάση την οποία συμμερίζομαι. Και ως εισηγήτρια είμαι αισιόδοξη για το ότι θα επιτύχουμε καλούς συμβιβασμούς και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για το λόγο αυτό θα προετοιμάσω τις ε, ακόλουθες συμβαστικές τροπολογίες. Πρώτον, στο άρθρο 3, διευκρίνηση και διεύρυνση των ε, προγραμματικών στόχων. Δεύτερον, διασάφηση των στόχων σχετικά με την ε, υπολογιστική υψηλού επίπεδου στο άρθρο 3. Έπειτα, ε, τεχνητή νοημοσύνη άρθρο 5, όπου θα προτείνω και τροπολογίες για την δεοντολογία του προγράμματος αυτού στο άρθρο 5. Θεωρώ πως η πρόθεση της ε, τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται να συνοδεύεται και από ένα διοντολογικό πλαίσιο. Επίσης, άρθρο 6, κυβερνασφάλεια, και εκεί θα καταθέσω συμβαστικές τροπολογίες, καθώς και πρόταση για διεύρυνση του προγράμματος ε, που αναφέρει το άρθρο 7. Οι συμβαστικές τροπολογίες θα περιλαμβάνουν λεπτομερή αναφορά των κέντρων καινοτομία στο άρθρο 16. Επίσης, αναγνωρίζω πως ελάχιστες ήταν οι τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, σχετικά με, την, με τον περιορισμό της πρόσβασης σε τρίτες χώρες, ε, συμπεριλαμβανομένων και των ε, υποψήφιων προς ένταξη χωρών, θεωρώ πως ένα τέτοιο βήμα θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες και θα πλήξει σημαντικά την ε, συνεργασία μας με τις χώρες αυτές. Δεν θα βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Στον τομέα της κυβερνασφάλειας είναι προς το συμφέρον μας να συνεργαζόμαστε στενά με χώρες οι οποίες θα χρησιμοποιούν διαλειτουργικές υποδομές και λύσεις και θα πρέπει να αποφύγουμε τον προστατευτισμό και να εξάγουμε τεχνολογία προηγμένη στον τομέα της κυβερνασφάλειας. Αυτά προς το παρόν. Θα χαρώ πολύ για τη συνεργασία με τους συναδέλφους ε, και όπως είπα είμαι αισιόδοξη για τις ε, τροπολογίες. Νομίζω πως θα καταφέρουμε να βρούμε ε, συμβαστικές λύσεις εκτός από τις ελάχιστες έτσι κάπως εθνικιστικού χαρακτήρα τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο τώρα από τους συναδέρφους. Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το έργο της. Ευχαριστώ για το περιεχόμενο επίσης των τροπολογιών. Διαβάζοντας έτσι για πρώτη φορά τις ε, τροπολογίες βλέπουμε ότι στηρίζουν το πρόγραμμα και υπογραμμίζουν διάφορα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για τον παρέτερο προβληματισμό σας. Από τη στιγμή που έχουμε περιορισμένο προπολογισμό. Και λέω περιορισμένο γιατί αν συγκρίνεται αυτά που προτείνουμε για το πρόγραμμα αυτό και αυτά τα οποία δαπανά η Ευρώπη συνολικά για αυτές τις σημαντικές ικανότητες, τεχνητή νοημοσύνη, ε, κυβερνοχώρο κτλ. Με τη σύγκριση αυτή δηλαδή διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μικρή επένδυση. Είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τα χρήματα αυτά για να οικοδομήσουμε τις ικανότητες ε, που χρειάζονται για να λειτουργήσουν τα προγράμματα. Και θα έπρεπε να προσέξουμε πώς δαπανούνται τα χρήματα. Για παράδειγμα, παράδειγμα από τις δεξιότητες. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα και το πρόγραμμα αυτό δεν λέω ότι θα λύσει όλα τα ζητήματα, χρειάζονται και άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Χρειάζεται συνεισφορά από τις χώρες μέλη. Αλλά επικεντρωνόμαστε εδώ κυρίως στο χτίσιμο δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ε, κόμβη ψηφιακής τεχνολογίας τώρα. Αυτή η ιδέα των ε, κόμβων τεχνολογίας θα παίξει σημαντικό ρόλο στις ικανότητες αυτές να είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες, αλλά κυρίως για τις χώρες και τις περιφέρειες εκείνες που δεν έχουν ακόμα επωφεληθεί τόσο πολύ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια απευθείας. αφορά τη συμμετοχή των τρίτων χωρών. Δίνουμε βέβαια μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή Αυτονομία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα για τρίτες χώρες τελικά να συμμετάσχουν. Φυσικά υπό προϋποθέσεις, υπό όρους ανάλογα με τις συμφωνίες που έχουμε με τρίτες χώρες και βέβαια βάσει διαφόρων ρητρών ασφάλειας. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υποφεληθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συμμετοχή τρίτων χωρών, γιατί η δικιά τους γνώση και ικανότητα μπορεί να βοηθήσει. Με αυτά τα σχόλια λοιπόν μπορώ να ολοκληρώσω. Πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε και θα καταλήξουμε σε ένα καλό σεβασμό και καλό πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Άλλος κανεί θέλει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκέπαρτ. Θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο ίσως δεν ταιριάζει σε αυτό το πρόγραμμα, όμως το θεωρώ αρκετά σημαντικό. Οι δεξιότητες, τις οποίες αναφέρουμε συχνά τελευταία, Χθε άκουσα μία παρουσίαση από έναν ερευνητή στον τομέα αυτών ο οποίος έλεγε ότι τα παιδιά του στο σχολείο δεν ε, μαθαίνουν καμία δεξιότητα όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα γενικότερα. Και νομίζω πως αυτό είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε μεγάλες ελλείψεις. Η ψηφιοποίηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να ενισχυθεί, όμως ε, χρειάζεται και τα παιδιά μας να μάθουν πώς να χειρίζονται τον, ε, τα μέσα, ε, πώς να μην πέφτουν σε παγίδες με ψευδείς ειδήσει και νομίζω πως ε, η παρουσίαση αυτή κατέστησε σαφές ότι τα παιδιά μας ε, ακόμα είναι σε αναλογικά, αν θέλετε, σχολεία, μαθαίνουν στον πίνακα, όχι με το ε, λάπτοπ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσουν και αυτές τις δεξιότητες. Νομίζω πως πρέπει να ενισχυθεί ο τομέας αυτός και σίγουρα η εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς δεν ε, μπορούμε και δεν πρέπει να ε, αναμειχθούμε, όμως ε, θα ήθελα να κάνω έκκληση στα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί από τις 9.30 και μετά θα πρέπει να φύγω, διότι ψηφίζουμε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και πρέπει να είμαι παρούσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο τώρα. Ο κύριος όμως Σάμιτ δεν είναι ακόμα εδώ. Η γραμματεία ίσως μπορεί να σας αναφέρει τις αποφάσεις που λήφθησαν χτες γύρω στις 6.30 στην συνάντηση των συντονιστών. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Την 10 Οκτωβρίου οι συντονιστές αποφάσισαν ακρόαση για ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και τα δικαιώματα των παιδιών διασυνοριακά. Επίσης, ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών όταν εφαρμόζουμε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να ζητήσει νομική γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 1 και του άρθρου 62 της συνθήκης στο άρθρο 114 για τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας για τα συγγραφικά δικαιώματα στα ψηφιακά. Αποφάσισαν επίσης να δεχτούν την πρόσκληση της Επιτροπής Αναφορών να έχουν ανταλλαγή απόψεων από κοινού με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια όσον αφορά την υπόθεση Αλμέγερ και επίσης την επόμενη Ολομέλεια να συζητηθεί. Και αυτή η συνάντηση θα γίνει στο Στρασβούργο, η έκτακτη. πρόεδρο. Ωραία. Περιμένουμε τον κύριο Ζάμιτ. Έχουμε εδώ βέβαια τον κύριο Σιέφκα. Αλλά έχω να σας κάνω δύο ανακοινώσει που θα συνδέσουν κατά κάποιο τρόπο τα ζητήματα αυτά. Έχουμε δύο επαιτίους σήμερα. Ο ένα δεν είναι εδώ ακόμα, οι άλλοι είναι εδώ. Κύριε Ντελβό, χρόνια πολλά. Έτσι δεν είναι. Αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ότι όλα αυτά θα χρησιμεύσουν σαν εισαγωγή για τον κύριο Ζιεύκα. Α, στο μεταξύ όμως ήρθε ο κύριο Τζάμιτ. Οπότε παρακαλώ κύριε Τζάμιτ έχετε το λόγο. Μόλις ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στην κυρία Ντελβό. Καταλαβαίνετε το κλίμα έτσι γίνεται πολύ ευχάριστο. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είχα μία συνάντηση με την Ταυτόχρονα θέλω να σας αναφέρω ότι τις ε, προηγούμενες εβδομάδες είχα διάφορες ε, συνεδριάσεις ε, με τα ενδιαφεραμένοι που εκπροσωπούν και τις πλατφόρμες και τους παρόχους για τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τον προτινόμενο κανονισμό. Επίσης, πήρα μέρος σε ένα φόρουμ που οργανώθηκε στη Μάλτα με τους stakeholders για το ίδιο θέμα. Οι τροπολογίες μου προσπαθούν να βρουν ισορροπία μεταξύ αυτών των διάφορων ενδιαφερομένων μερών τον θερεντικό για μένα ότι και οι εκπρόσωποι από τις πλατφόρμες αλλά και από τις επιχειρήσεις καλώς ορίζουν το σχέδιο γιατί, κανονισμού γιατί αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη για το πώς λειτουργεί η ενιαία αγορά σε ψηφιακό επίπεδο και πρέπει να προωθήσουμε την διαφάνεια και την ε, ισότητα. Θα αναφερθώ σε διάφορα θέματα. Διάφορες ε, επιχειρήσεις μας ε, ε, κοινοποίησαν τις ανησυχίε τους σε σχέση με το θέμα της ε, κατάταξης. Ε, δεν... Θα ξεχάσω ότι μου έδωσαν και κάποιες αποδείξεις και μας έδειξαν ότι κάποιες πλατφόρμες Προφανώς, ε, αλλά μόνο αν το ψάξει κανείς, δίνουν προτίμηση σε προϊόντα και υπηρεσίες ε, που παρέχουν ε, αυτές οι ίδιες στην αγορά ή δίνουν προτίμηση σε κάποιους προτινόμενους παρόχους υπηρεσιών που, ε, επιχειρήσεων με τις οποίες έχουν συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες. Επομένως, είναι ζωτικό να έχουμε διαφάνεια για τα κριτήρια που καθορίζουν την κατάταξη. Ταυτόχρονα δέχτηκα το επιχείρημα που έγινε από τον εκπρόσωπο των πλατφορμών ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ολόκληρους τους αλγορίθμους γιατί θεωρούν ότι είναι εμπορικό απόρριτο και επίσης θεωρούν ότι αυτό μπορούν να δώσουν ε, εκ των προτέρων, ε, ανταγωνίζονται τις υπόλοιπες πλατφόρμες, αλλά αν δοθούν ε, και οι αλγόριθμοι, τότε οι επιχειρήσεις ε, μπορούν να εργαστούν επί των επιτελεσμάτων ε, δρώντας επί συγκεκριμένων κριτηρίων επί του αλγορίθμου. Χρειαζόμαστε λοιπόν γενικά κριτήρια κατάταξης, αλλά όχι τους συγκεκριμένους αλγόριθμους. Οι τροπολογίες ε, που έχουν παρουσιαστεί προσπαθούν να κάνουν μια διάκριση μεταξύ των ίδιων των συναλλαγών, και της έναρξης μιας συναλλαγής. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται να αγοράσει ένα προϊόν. Εγώ, το χάρη, θα ήθελα να αγοράσω, το χάρη, έναν υπολογιστή, μια τηλεόραση, ένα αυτοκίνητο και κάνω έρευνες και πάω στις ιστοσελίδες των διάφορων προϊόντων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχω ξεκινήσει μία συναλλαγή για να αγοράσω. Πώς αυτή η έρευνα στη συνέχεια, λοιπόν, ε, να σημαίνει ότι θα πρέπει να ολοκληρώσω τη συναλλαγή. Από την άλλη υπάρχει μια διαδικασία, οπότε μπορείς να καθορίσεις ότι υπάρχει έναρξη της συναλλαγής και όταν υπάρχει τέτοια έναρξη της συναλλαγής, τότε θα πρέπει να προστατεύσουμε την πλατφόρμα. Ένα άλλο θέμα που ανέκυψε στις διαβουλεύσεις αφορά την απέτηση ε, παροχής εσωτερικών μηχανισμών ε, ένωμης προστασίας ε, και διαμεσολάβησης. Νομίζω ότι εδώ θα ήταν σόφρο να δεχτούμε το επιχείρημα ότι μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε ένα κατόφλι με χάρη ε, του αριθμού των μοναδικών ουσιαστικά των μοναδικών συναλλαγών, γιατί τότε δεν θα πρέπει ε, να επιβάλλεται στις μικρές πλατφόρμες να μας παρουσιάσουν τον εσωτερικό τους μηχανισμό. Οι μεγάλες πλατφόρμες μπορούν να το κάνουν και πρέπει να έχουν φυσικά άμεση σχέση με τους ε, παρόχους ε, των... Αλλά αν επιβάλλουμε στους μικρούς, αυτά που θέλουμε να επιβάλλουμε στους μεγάλους, ε, τότε θα τους βλάψουμε και δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Φυσικά υπάρχουν κάποια θεμελιώδη κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν σε όλους. Και το λέω αυτό γιατί κάποιες ε, πλατφόρμες ε, μας είπαν το εξή: ότι ε, αυτός ο κανονισμός τελικά θα ισχύει μόνο για τους μεγάλους. Και εγώ είπα αυτό πηγαίνει πολύ μακριά. Επίσης είχαμε παρουσιάσεις για όλο το θέμα της διαμεσολάβησης. Πιστεύω ότι σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι επιθυμητό διαμεσολάβηση, αλλά όχι υποχρεωτικό. Η διατύπωση της Κομισιόν ήδη ενέχει ότι είναι κούσιο, αλλά μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε περισσότερο. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο χρήστης ε, μπορεί να, ο επιχειρηματικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δικαστικές, τη δικαστική οδό πέραν της διαμεσολάβησης. Αυτά είναι όσοι ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ τους κυρίους ε, ε, Μπάγνους και Ντόρματσοκ για την ε, βοήθειά τους. Χθες το βράδυ με βοήθησαν πάρα πολύ και θέλω να τονίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι στις 24 Οκτωβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. κυρία Ρέτα. Ευχαριστώ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη εκ των προτέρων, γιατί θα πρέπει να φύγω για τι ψηφοφορίε αμέσω μετά την παρέμβασή μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για εξαιρετικό σχέδιο γνωμοδότηση. Νομίζω πράγματι βρίσκει μια ισορροπία μεταξύ των πλατφορμών και των επιχειρήσεων και έχει και προσθέμενη αξία για του καταναλωτέ που χρησιμοποιούν αυτέ τι πλατφόρμε αλλά και τι επιχειρήσει. Μπορώ να κατανοήσω τη λογική να κάνετε μία διάκριση μεταξύ της έναρξης μιας συναλλαγής και της υλοποίησης της συναλλαγής και νομίζω ότι στη γνωμοδότηση περίπτωση χάρη μια ιστοσελίδα σύγκριση τιμών δεν θεωρείται πλέον πλατφόρμα. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά κατόπιν νομίζω ότι πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι όντω ε, θεωρείται μηχανή αναζήτηση, γιατί θα πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο για να μην δημιουργήσουμε νομικό κενό. Επίσης είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε και την φωνητική βοήθεια στον ορισμό της μηχανής αναζήτησης. Επίσης συμφωνώ με την ιδέα να πούμε ότι αν κάποιος έχει αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς μια περίοδο πρώτερη ενημέρωσης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις καθόλου. Απλώ ε, να διασφαλίσουμε ότι ισχύει η περίοδο κοινοποίηση ορισμένε περιπτώσεις μια πλατφόρμα μονομερό θα μπορούσε να αλλάξει τι προποθέσει και του όρου, χωρί να έχει καθόλου περιδοκινοποίηση. Αυτό με προβληματίζει γιατί φοβάμαι πολύ συχνά οι πλατφόρμες θα χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι πρέπει να προστατεύσουν την πλατφόρμα του ή κάτι τέτοιο. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ασφαλιστικέ ασφαλιστικές Σε Ό,τι αφορά τα κριτήρια κατάταξη όλοι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι διαφανές το πώς λειτουργεί η έρευνα ή η κατάταξη. Δεν θέλουμε να δημοσιεύονται οι αλγόριθμοι και πιστεύω ότι το σχέδιο γραμματότησης δηλώνει ακριβώς αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν σε κατάχρηση να αποκαλυφθούν, αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη είναι το ερώτημα. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να υπάρχει ένας κίνδυνος ότι μπορεί να το αναφέρει αυτό κάποιο επιχείρημα, ενώ δεν θα ισχύει. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε για να μην δημιουργήσουμε νομικό κενό. Ανέφερα και το θέμα της προστασίας των δομένων. Στην γνωμοδότηση το καλωσορίζω. Νομίζω ότι θα είναι καλό να αναφερθούμε στο γενικό κανονισμό προστασίας των δομένων παρά στις πολιτικές εμπιστευτικότητας των πλατφορμών. Καλωσορίζω πάρα πολύ την προσθήκη ότι οι να τεθεί λήξη να καταγγελθεί ένας λογαριασμός ή μια σύμβαση θα πρέπει να είναι μόνο διαφανής αλλά και αναλογικές. Νομίζω ότι ουσιαστικά εδώ τονίζεται το κριτήριο της δικαιοσύνης στην έκθεση αυτή. Επίσης, το γιατί να συμπεριλαμβάνονται κάποιες υποχρεώσεις παροχής ε, πληροφοριών ε, προς τις ε, πλατφόρμες από τις εγχειρήσεις. Εδώ βασιζόμαστε στον κανονισμό μνημπούς όπου επαιτείται οι πλατφόρμες να δίνουν κάποιες πληροφορίες στους καταναλωτές που αφορούν τις επιχειρήσει. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν αυτές τις πληροφορίες, επομένως αυτό χρησιμεύει ως προσθήκη. Δεν συμφωνώ με το να αποδυναμώσουμε τις υποχρεώσεις διαφάνειας των πλατφορμών σε σχέση με το εσωτερικό του σύστημα καταγγελιών έτσι λοιπόν, ίσως θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε λίγο περισσότερο σε ποιο βαθμό οι διάφορες πλατφόρμες μπορούν να έχουν αυτά τα συστήματα. Νομίζω όμως ότι η διαφάνεια των συστημάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ενίοτε οι ανταγωνιστές χρησιμοποιούν, παραδείγματο χάρη, κάποιες κοινοποίησεις που στέλνονται στις πλατφόρμες ως μέσος του ανταγωνισμού. Θέλουν δηλαδή να αφαιρεθούν οι καταχωρήσει των ανταγωνιστών. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει εντοπίσει η Κομισιόν και στη μελέτη αντικτύπου. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο να έχουμε μεγάλη διαφάνεια σε ό,τι αφορά το σύστημα καταγγελία και σε ό,τι αφορά και τι κοινοποίησει που στέλνονται από του ανταγωνιστέ και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν καταχρήσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και ασφαλιστικέ δικλείδε στο σύστημα διαμεσολάβηση. Έτσι λοιπόν, αν παραδείγματο χάρη ένα χρήστη ε, προβαίνει σε κατάχρηση του μηχανισμού, τότε θα πρέπει να έχει υψηλότερο οικονομικό άχθο. Και σε ό,τι αφορά τώρα τη συλλογική ένωμη προστασία, νομίζω ότι είναι καλό να βάλουμε κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι θα εξακολουθεί να λειτουργεί η ένωμη προστασία στην πράξη, η προσφυγική δικαιοσύνη, γιατί είναι μια μεγάλη καινοτομία τη πρόταση. Τέλο, καλωσορίζω τα όσα υπόθηκαν από τον εισηγητή στη ρήτρα αναθεώρηση, ε, δηλαδή να διερευνήσουμε το αν μπορεί να καλύπτει ο κανονισμό και τα συστήματα ε, λειτουργία ε, και να υπάρχει και πιθανή απαγόρευση θέμη των ε, εμπορικών πρακτικών. Πρέπει να διερευνήσουμε περαιτέρω αυτή την ιδέα. Ανυπομονώ λοιπόν να συνεργαστώ μαζί σα για την γνωμοδότηση αυτή και Καθώς εγώ παρακολουθώ το φάκελο και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ θέλω να διασφαλίσω ότι θα είναι ισχυρή η φωνή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων στη διαδικασία αυτή και θα προωθήσει πολλά από αυτά τα σημαντικά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρέντα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ και σύντομα γιατί αρχίζουμε να καθυστερούμε ενώ είμαστε στην αρχή ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή και την Επιτροπή σας για τη γνωμοδότηση αυτή και για την δυνατότητα που μας δίνετε να πούμε και εμείς δύο λόγια. Σύντομα. Ευχαριστούμε για το έργο σας και συμφωνούμε με πολλά από τα στοιχεία της γνωμοδότησης αυτής. Κυρίως βέβαια ότι η βασική φιλοσοφία της πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται κατανοητή και συμφωνεί και η δικιά σας Επιτροπή. Σε δύο σημεία θα σταθώ που πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν προχωρήσετε με τις τροπολογίες. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρόκειται για μια προσέγγιση σε δύο στάδια και αυτό πρέπει να το τονίσουμε για να το υπογραμμίσουμε και το υπογραμμίσαμε και στην ε, μελέτη αντικτύπου εμείς δεν θα αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα από την αρχή. Θα δημιουργήσουμε μια διαδικασία σε δύο στάδια, οπότε πρώτα θα δούμε πού υπάρχουν ε, αποδείξεις και είναι κατάφορο ότι υπάρχουν συστημικά ζητήματα με εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα συγκεντρώσουν στοιχεία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλο και περισσότερο ώστε να ετοιμάσουμε την αναθεώρηση. Κάτι το οποίο αναφέρεται και σε κάποιες τροπολογίες που προτείνατε. Το δεύτερο σχόλιο μου, και θα σταματήσω μετά, είναι προσοχή σε ένα μικρό στοιχείο που δεν είχε αναφερθεί νωρίτερα, που προτείνει στην τροπολογία 32 ο εισηγητής να πάμε πέρα από τον ε, κανονισμό, δηλαδή ότι οι χώρες μέλη μπορούν να πάνε πέρα από τον κανονισμό. Μην ξεχνάμε ότι η νομική βάση είναι η εσωτερική αγορά. Και άρα πρέπει να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατόν βαθμός εναρμόνισης. Αυτό ήθελα να σας πω, να το έχετε υπόψη σας πριν καταλήξετε σε αποφάσεις. Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ πολύ για το καλό αυτό σχέδιο γνωμοδότησης και είμαστε στη διάθεσή σας για τη συνέχεια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σύντομος. Εσείς, ε, συγητής, κύριε Σάμιτ, θέλετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέρφους που πήραν το λόγο και από αυτά που άκουσα βγάζω το συμπέρασμα ότι θα μπορέσουμε πολύ εύκολα να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε στην τελική έκθεση. Να απαντήσω στα σχόλια. Για τις μηχανές έρευνας, ναι, πράγματι δεν είχα, όπως καταλαβαίνετε, χρόνο να τα βάλω όλα σε αυτό το κείμενο. Ναι, η φωνή, ναι, να συμπεριλαμβάνεται, συμφωνώ. Τώρα όλο το θέμα, το κατά πόσο θα δεχτούμε παρόχους μερικές φορές... Ε, να ξέρετε ότι κάποιοι έχουν ε, αποδείξει και μας έχουν πείσει ότι πρέπει κανείς να πηγαίνει γρήγορα. Δηλαδή, όταν υπάρχει απάτη, φαίνεται να υπάρχει η απάτη ή όταν δεν υπάρχει εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ένα εστιατόριο υποτίθεται ότι είχε συναλλαγή, αλλά δεν ήταν. Δηλαδή, είχε καταφέρει αυτός να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν εστιατόριο. Με την κατάταξη, με όλα εκεί δεν μπορείς να περιμένεις, πρέπει αμέσως να δράσεις. Άρα πρέπει να το καταλάβουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις θα πρέπει να δρούμε γρήγορα. Συμφωνούμε με αυτά που είπατε για τους αλγόριθμους, με την προστασία δεδομένων, μπορούμε να απευθυνθούμε και στον υπόπτη δεδομένων. Συμφωνώ και με την αναλλαγικότητα και από αυτού υπάρχουν τροπολογίες. Ε, συστήματα εσωτερικών προσφυγών πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να προστατεύουμε τους μικρότερους παίκτες. Υπάρχουν δηλαδή επίπεδα διαφάνειας που ισχύουν για όλους τους παρόχους πλατφόρμων. Συμφωνώ επίσης για τις συλλογικέ ε, πανορθώσεις. Οι ρήτρε ασφάλεια που ανέφερα εγώ είναι για να διασφαλίσουμε ότι αυτό ο μηχανισμός συλλογική διόρθωση δεν είναι για να βγει κανείς κερδισμένος. Το λέω πολλές φορές στις συναντήσεις μου, με κάθε σεβασμό βέβαια για την Αμερική, αναφέρομαι στο αμερικανικό νομικό σύστημα, όπου είναι γνωστό ότι οι δικηγόροι ε, τα κυνηγούν διάφορες υποθέσεις, κυνηγούν ας πούμε τα ασθενοφόρα για να βρούνε ποιο είναι μέσα και μετά πάνε και τον πλησιάζουν και του λένε να τον υποστηρίξουν για να βγάλουν χρήμα. Πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα πράγματι πηγαίνουν στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από κάποιο πρόβλημα και όχι στις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν. και στην ΙΜΚΟ φαντάζομαι έχουν εκατοντάδες τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο να συγκλίνουν οι απόψεις των δύο επιτροπών. Όσον αφορά τώρα τη συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων και το παρατηρητήριο, συμφωνώ. Και μάλιστα προτείνω μετά από δύο χρόνια να είναι η περίοδος αναθεώρησης και όχι μετά από τρία χρόνια όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και θέλουμε να έχουμε feedback όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και τέλος, κατά πόσο οι χώρες μέλη θα μπορούν ή όχι να πάνε πιο μακριά ακόμα. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι δύσκολο να δει το φως ο κανονισμός αυτός, αν δεν το επιτρέψουμε αυτό. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποιες χώρες έχουν τους δικούς τους εθνικούς νόμους για αυτό το ίδιο ζήτημα. Υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία πολλές φορές όπου δεχόμαστε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο το οποίο πρέπει να πετύχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά λέμε ότι αν κάποιες χώρες θέλουν να προσφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα ε, προστασίας, μπορούν, εκτός βέβαια αν πλήττονται οι κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας κλπ. Αν δεν το επιτρέψουμε αυτό, είναι σαν να προσπαθούμε ευθύ εξ αρχής να βρεθούμε σε σύγκρουση με χώρες όπως η Γαλλία, η οποία έχει πολύ καλούς νόμους γι' αυτά να έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά να λέμε ότι αν κάποιος θέλει να πάει πιο μακριά ακόμα, να το κάνει, αρκεί να μην πλήττονται οι κανόνες ελεύθερης κυκλοφορίας και ανταγωνισμού. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας, αγαπητέ συνάδελφε. Χωρίς άλλα σχόλια, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξη, σημείο 30. Ο κύριος Ζιέφκα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα θα συζητήσουμε τις τροπολογίες που κατατέθηκαν για την έκθεσή μου και επιτρέψτε μου να αρχίσω με ένα γενικότερο σχόλιο. Όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες μας για την έκθεση, για την πρόταση της Επιτροπής, οι αρχικές αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές. διότι η πρόταση αφορούσε κάτι που θα βελτίωνε κατά πολύ τη λειτουργία των εταιριών στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τότε είχαμε συμφωνήσει ότι αυτές οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν και ήταν κατάλληλες για το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι καθημερινότητα πλέον και εκεί λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες και διοικητικέ και δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε και οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται και ψηφιακά και να κάνουν διάφορα επιγραμμικά. Επίσης, για τους νέους, ε, το ψηφιακό περιβάλλον είναι το φυσικό ενδιέτημά τους, αν θέλετε. Γι' αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση που κατατέθηκαν τέτοιες τροπολογίες και τόσες πολλές, 256. Τις διάβασα και παρατηρώ ότι ασκείται έντονη κριτική στην πρόταση της Επιτροπής. Ή έστω προσπαθείτε να περιορίσετε τα μέσα που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Προτού λοιπόν περάσω στις τροπολογίες, θα απαντήσω σε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, όπως ε, είπαμε και στην αρχή, Θέλουμε πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό, φιλικό προς το χρήστη τρόπο καταχώρησης εταιριών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά της ε, Ευρώπης. Πώς θα το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα καταχώρησης επιγραμμικά, χωρίς να χρειαστεί κάποιος ε, εκπρόσωπος να πάει αυτοπροσώπως στις ε, αρμόδιες υπηρεσίες να συμπληρώνει έντυπα. Καταργώντας όλα αυτά και επιτρέποντας ε, να γίνεται η διαδικασία μέσω του διαδικτύου σύντομα και χωρίς ε, πρόσθετο φόρτο. Αν η απάντηση σε αυτήν την απλή ερώτηση είναι ναι, τότε θα ήθελα να πω ότι ο πιο εύκολος και σύντομος τρόπος είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. διότι η πρόταση αυτή επιτρέπει την δυνατότητα αυτή καταχώρησης ηλεκτρονικά μίας ε, εταιρείας χωρί... εναρμονίζοντας το ουσιαστικό δίκαιο, χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους κανόνες που χρησιμοποιούν σήμερα τα κράτη-μέλη. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση ο όγκος των ε, τροπολογίων και το περιεχόμενό τους. Γιατί από αυτές φαίνεται ότι αυτή η αρχικά θετική προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια κατάσταση διαφορετική όπου οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ε, ανοίγουν υποκαταστήματα ή να ε, συστήνουν μια εταιρεία σε κάποιο άλλο κράτος μέλος. Μπορούμε να χωρίσουμε τις τροπολογίες σε τρεις κατηγορίες. Οι πρώτες ε, αφορούν το πεδίο εφαρμογή, η δεύτερη την καταχώρηση των ίδιων των εταιριών και τρίτον τα υποκαταστήματα σε τρίτες χώρες, ίσως και μια τέταρτη ομάδα τροπολογιών που αφορά ε, τις ε, πληροφορίες που θα καταχωρούνται στα Μητρώα. Νομίζω καταρχάς ότι ω προ το πεδίο εφαρμογή, όσο μεγαλύτερο είναι τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ίσως να μην είναι ορατό από την αρχή, όμως νομίζω ότι η απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο θα έχει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και θα αλλάξει τον τρόπο που ε, λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αυτό θα φανεί και στην αγορά. Βέβαια, κατανοώ ορισμένες ανησυχίες που εκφράστηκαν διότι το πεδίο εφαρμογής είναι αρκετά ευρύ και καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχουν διάφορες μορφές εταιριών Καταλαβαίνω επίσης και τις ε, παραδόσεις κάθε χώρας που έχουν να κάνουν με την καταχώρηση, με την εποπτεία των εταιρεών κτλ. Όμως αν θέλουμε να εξυγχρονιστούμε και να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα επιφέρει προστιθέμενη αξία. Ένα σύστημα το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όμως περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογή, θα περιοριστούν και οι μορφές των εταιριών που μπορούν να καταχωρηθούν. Ποιες εταιρείε δηλαδή, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, θα είναι πολύ στενό το πεδίο εφαρμογή και στη συνέχεια αυτό θα έχει και επιπτώσεις. Αν επιτρέψουμε και στα νομικά πρόσωπα να κάνουν αυτή την επιγραμμική καταχώρηση, τότε κινδυνεύουν να εμφανιστούν διάφορες ε, ύποπτες ε, περιστάσεις, εταιρείες βιτρίνες κτλ. Χρειάζονται πληροφορίες βέβαια, να δούμε τι είναι αυτές οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Ε, στα νομικά πρόσωπα όμως αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ πιο εύκολο να ελεγχθούν παρά σε ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο ενδεχομένω δεν ξέρει κανείς ε, τι έκανε στο παρελθόν. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να καταχωρήσει μια εταιρεία και στη συνέχεια να την πουλήσει όποιον θέλει, σε ένα νομικό πρόσωπο. Παρακάμπτοντας έτσι το μηχανισμό αυτό. Όμως, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι υπάρχει γενικότερη υποψία ότι όλοι θέλουν να εξαπατήσουν. Η νομοθεσία όμως που θέλουμε να περάσουμε δεν ε, αφορά τους απατεώνες, αλλά τους ε, ειλικρινείς επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν καλόπιστα να δραστηριοποιηθούν με τις επιχειρήσεις τους. Σε περίπτωση απάτης υπάρχουν οι απαραίτητοι φυστάμενοι μηχανισμοί που αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν οι αμφιβολίες που ίσως έχετε και αναφέρονται σε αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεν ευσταθούν και τόσο πολύ. Τώρα σε ό,τι αφορά την καταχώρηση. Το σύστημα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται στις ίδιες εθνικές αρχές οι οποίες ισχύουν όταν γίνεται καταχώρηση μιας εταιρείας με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, με τα έγγραφα πρέπει κανείς να καταθέσει κτλ. Ο ετών θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της χώρας. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν θα χρειαστεί να πάνε οι ίδιοι προσώπο σε κάποια υπηρεσία, σε ένα γραφείο, αλλά μπορούν να το κάνουν από το διαδίκτυο. Γι' αυτό νομίζω πως θα έπρεπε να δώσουμε έμφαση σε αυτήν την πτυχή της οδηγίας, δηλαδή το στοιχείο της αμοιβαία εμπιστοσύνη. για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ήδη υπάρχουν αυτές οι δομές, υπάρχει το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. υπάρχουν ηλεκτρονικές συναλλαγές στην ενιαία αγορά και τα συστήματα αυτά μια χαρά φαίνεται πως λειτουργούν. Τώρα, κάποιες από τις τροπολογίες έχουν στόχο να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσει οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σε κάποια κρατημέλη. Γι' αυτό αν γίνουν δεκτές θα επιδεινώσουν την νομοθεσία, ιδιαίτερα σε κάποια κράτη-μέλη που ήδη εφαρμόζουν την ηλεκτρονική καταχώρηση εταιριών. Στην πρόταση της Επιτροπής τα κράτη-μέλη είναι αυτά που υποχρεούνται να παράσχουν έντυπα για, τις, ε, για την καταχώρηση εταιριών ή θηγατρικών. Ο κύριος Ρόντε από τους φιλελεύθερους κατέθεσε μία τροπολογία η οποία δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να δημιουργήσει πρότυπα έντυπα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να μπορεί, ε, τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να καταχωρήσει μια εταιρεία, μια θηγατρική σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μπορεί να μας ενημερώσει για το κατά πόσο εφικτή είναι μια τέτοια πρόταση. Μετά, η καταχώρηση μιας εταιρεία. Θα προστατεύεται από απάτη πώς. απαγορεύοντας κάποιο πρόσωπο να κρατά ε, διευθυντική θέση σε ένα άλλο κράτος μέλος. Κάτι τέτοιο ήδη υπάρχει. Αυτή η απαγόρευση εκδίδεται από μια εθνική αρχή με βάση κανόνες μίας χώρας που δεν ισχύουν σε μια άλλη. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή προσεγγίζοντας ε, από αυτήν την κατεύθυνση το θέμα. Νομίζω πως χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μητρό όπου θα αναφέρονται τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει αυτή η απαγόρευση και θα είναι ανοιχτό σε όλους τους ετούντες. Ε, τώρα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει πολλές φορές και σε πολλές επιτροπές. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μητρό, θα πρέπει να περιορίσουμε την πρόσβαση, έτσι ώστε η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένες ε, οντότητες. Επίσης, τέλος, να αναφερθώ στην πρόσβαση στην πληροφορία. Φυσικά και θέλουμε την ε, μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι αυτή η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία επιφέρει και κόστος για τις αρμόδιες αρχές. Τα τέλη που καταβάλουν όσοι θέλουν να καταχωρήσουν μια εταιρεία δεν καλύπτουν το κόστος λειτουργίας αυτού του Μητρώου. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο να εξισορροπήσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτά λοιπόν από μένα. Αυτά είχα να πω. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τα δικό σας σχόλια και τα σχόλια της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Συγητή. Η κυρία Κούτελα έχει το λόγο. Θα ζητήσω στους επόμενους ομιλητές να μην με ακρηγορήσουν γιατί ήδη έχουμε συσσωρεύσει καθυστέρηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ζεύσκα για το έργο του, για αυτό το σημαντικό φάκελο. Καταρχήν θέλω να μιλήσω γενικότερα για την οδηγία αυτή. και ως μέρος όλης της δεσμής μέτρων για το εταιρικό δίκαιο. Όταν σας ακούω να μιλάτε για αυτό το σημαντικό φάκελο, κάπως μπερδεύομαι, γιατί νιώθω ότι είστε κάπως αμυντικός απέναντι στην βελτίωση της πρότασης ε, βάσει των τροπολογιών που είδατε, αλλά πρέπει να σας ε, διαβεβαιώσω για να ξεκινήσουμε από αυτό ότι η πρόταση δεν είναι κάτι που εγώ επικρίνω ως ε, ένας ε, δρόμος προς το μέλλον, ούτε η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές. Ξεκάθαρα είναι μια σημαντική πρόταση, ζούμε στην ψηφιακή εποχή, βλέπουμε την ανάγκη να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, βλέπουμε ότι η Κομισιόν κάνει σημαντική δουλειά προσπαθώντας να αναπτύξει και να βελτιώσει περαιτέρω την εσωτερική αγορά στους καιρούς που ζούμε, όταν βλέπουμε ότι θα πρέπει να εργαστούμε διασυνοριακά και θα πρέπει να απλωστεύσουμε το πώς δουλεύουμε στο διαδίκτυο. Βέβαια δεν θέλω να τα τονίσω αυτά γιατί αυτά είναι εντός της πρότασης. Πρέπει να υπογραμμίσω το πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες ό,τι αφορά την πρόταση αυτή. Και αυτό το κάνω φιλικά. Και η ομάδα μου το κάνει φιλικά. Γιατί όπως υπόθηκε, ο εχθρός ε, θα είναι σιωπηρός όταν ε, θα έχεις προβλήματα, αλλά ο φίλος θα μιλήσει και θα σε βοηθήσει, θα σου μιλήσει ειλικρινά και θα προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάστασή σου. Και εγώ αυτό σκοπεύω να κάνω. Η πρόταση αυτή πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη που έχουν ένα καλό σύστημα ε, που αφορά την ορθή απονομή της δικαιοσύνης να συνεχίσουν να προσφέρουν δικλείδες ασφαλείας στους κυρίους που ζούμε όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν καταχρήσεις σε ό,τι αφορά την διασυνοριακή συμπεριφορά των εταιριών. Πιστεύω ότι προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα μητρώα των επιχειρήσεων είναι αξιόπιστα και ότι η οδηγία θα τις βοηθήσει να είναι επικαιροποιημένες με το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ζητήσουν φυσική παρουσία σε ευρύτερο πλαίσιο, πέρα από το αν υπάρχει πραγματική υποψία απάτης, αν αυτό αιτιολογείται από κάποιο λόγο δημοσίου συμφέροντος, παραδείγματος χάρη, όπως η καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Η Κομισιόν στην πρόταση μας ε, λέει ότι ο στόχος ε, με την οδηγία αυτή δεν είναι να ερμονίσει ουσιαστικές απαιτήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με τις εταιρείε γραμματοκιβωτίου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιούμε τον κίνδυνο ε, της βαρδιοφυγής, της νομοποίησης παράδειγμας εισόδων και της ψευδούς απασχόλησης αν αυτή η οδηγία δεν έχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ότι ένας καλός συμβιβασμός ό,τι αφορά την ενδυνάμιση των ρόλων ε, όπως ε, θα έχουν οι αρμοδίες αρχές στα δικαστήρια ε, και άλλοι φορείς διαφύλαξης του νόμου θα λειτουργούν γιατί βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο έχουμε προβλήματα με την απάτη και ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη υποφέρουν από κάποιες εταιρείε που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, που δεν πληρώνουν τους φόρους, παραδείγματο χάρη. Το σύστημα πρόνοιας το χρειάζεται αυτό. Επομένως, ε, είναι πολύ σημαντικό από πολιτική σκοπιά, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Στο παρελθόν συζητήσαμε την απέτηση να έχουμε δωρεάν πληροφορίες για τις ε, εταιρείες ε, που είναι στο σύστημα σε σχέση με το σύστημα διασύνδεσης μικρών επιχειρήσεων. Πολλοί έχουν καταθέσει τροπολογίες να αυξηθεί, να αυξηθούν πληροφορίες σε σχέση με τον αριθμό των απασχολουμένων και δυνάμει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και όχι μόνο όταν απαιτείται από την Εθνική Νομοθεσία όπως προτείνεται από την Κομισιόν. Αυτή η διαφάνεια επίσης θα βελτιώσει την πρόταση. Θέλω να πω εδώ ότι η περισσότερη διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση προωθεί την αμοιβαία εμπιστοσύνη, ενδυναμώνει το διάλογο, μας προσφέρει αξιόπιστα δεδομένα για την κατάσταση των επιχειρήσεων, αυξάνει την ευαισθησία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στους υπαλλήλους και τους επενδυτές. Επίσης προωθεί την εμπλοκή των υπαλλήλων στο μέλλον της εταιρείας και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα. Περισσότερες δωρεάν πληροφορίες ε, είναι κάτι θετικό για όλους, για τις εταιρείες, ε, τους εργαζομένους και την ανάπτυξη των εταιριών. Πρέπει να την προωθήσουμε λοιπόν. Τέλος, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι το ψηφιακό εργαλείο είναι μία από τις δύο νομοθετικές προτάσεις εντός της δεσμημέτρων για το εταιρικό δίκαιο και θα πρέπει αυτά να συμβαδίζουν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμβαδίζουν όντως αυτά και να διασφαλίσουμε ότι ε, ουσιαστικά αυτά λειτουργούν ανάλογα και με το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ κύριο Σωτόφσκι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω ότι το ECR υποστηρίζει τη θέση του εισηγητή και δεν βλέπουμε λόγους να υποβάλουμε τροπολογίες. Συμφωνούμε με όλα τα μέτρα που προτείνονται διευκολύνουν ε, το να συσταθεί μια εταιρεία μέσω του διαδικτύου. Όμως αυτό το επιγραμμικό εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευρέως ε, για την εγγραφή στο Μητρό των εταιριών. Τώρα, το να περιορίσουμε το πεδίο εφημερογή ε, δεν δικαιολογείται γιατί δεν θα έχει αντίκτυπο η πρόταση στο να περιορίσουμε το κόστος. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν τον εισηγητή στο περαιτέρω έργο του. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο σύντομος η Κομισιόν. Και επίσης έχετε την ίδια σύσταση κι εσείς, αν θέλετε, να τη λάβετε υπόψη. Σας ευχαριστώ που δεν θα με κρηγορήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα μια ερώτηση από τον εισηγητή προς την Κομισιόν σε σχέση με τα templates, ε, αυτά τα έντυπα, τα πρότυπα έντυπα αν μπορούν να ετοιμαστούν ε, από την Κομισιόν για να χρησιμοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πρόταση αναφερόμαστε σε εθνικά έντυπα, γιατί θέλουμε να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι δυνατό να εργαστούμε με ευρωπαϊκά τέτοια έντυπα, αλλά δεν θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σόφρον. Γιατί θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να χρησιμοποιηθούν γιατί δεν είναι αρμονισμένοι οι εθνικοί κανόνες. Θα ήταν λοιπόν πολύ πλοκό να προετοιμάσουμε αυτά τα έντυπα με τόσες διαφορετικές ε, επιλογές. Είναι δυνατό, αλλά είναι ιδιαίτερα πολύ πλοκό. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι έχουμε ένα feedback ότι τα εθνικά έντυπα ε, λειτουργούν καλύτερα, ακόμη και στις περιπτώσεις ε, που εμπλέκονται και άλλοι επαγγελματίε όπως οι συμβολογράφοι. Θεωρούμε ότι αυξάνουν την ασφάλεια δικαίου και επιταχύνουν και τη διαδικασία εγγραφής. Επομένως, ε, θεωρούμε ότι το να προσφέρουμε ε, τα template αυτά να εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη είναι η καλύτερη λύση. Και το δεύτερο σχολείο μου έχει, μετά να τονίσουμε ότι η Κομισιόν συμφωνεί με την ανάλυση του εισηγητή σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή. Πιστεύουμε ότι ο περιορισμό του πεδίου εφαρμογή και το να μην επιτρέπουμε την εγγραφή νομικά πρόσωπα πραγματικά θα φερούσε πολύ μεγάλη αξία από την πρόταση. Θεωρούμε ότι θα ήταν ε, ουσιαστικά εισαγωγή διακρίσεων, να μην επιτρέψουμε σε εταιρείε, μάλλον σε ένα νομικό πρόσωπο, να ιδρύσει θηγατρικέ σε άλλε χώρε. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε οποιαδήποτε τεχνική βοήθεια χρειάζεται για να επιλύθουν τα πρακτικά προβλήματα. Όμως ελπίζουμε ε, ότι θα ακολουθηθεί η γραμμή του συγητή σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι αν δεν ε, υπάρχουν πιθανότητες τα νομικά πρόσωπα να ιδρύσουν θηγατρικές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα κράτη-μέλη θα έχουν τα δικά τους πρότυπα για το αν αυτό είναι δυνατόν ή όχι. Και αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για το θέμα της ασφάλειας δικαίου και θα μπορούσε να δώσει χώρο σε απάτες ή καταχρήσεις. Έτσι λοιπόν, Μας ε, ενδιαφέρει να υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές ε, δικλίδες και να αναγράφονται ξεκάθαρα στον Ευρωπαϊκό Νομοθέτημα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριο Ζεύκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την απάντηση στην ερώτηση. Αυτό ξεκαθαρίζει τα ερωτηματικά που είχα. Σας ευχαριστώ όλους. να πω και δύο λόγια για να κλείσουμε. Οτιδήποτε θέλει να συμβάλλει στη βελτίωση του κειμένου, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να καταπολεμηθούν οι κατακρίσει, έχει αντιμετωπιστεί από μένα με τη μεγαλύτερη κατανόηση. Φυσικά είμαι απολύτω υπέρ, όμω δεν συμφωνώ με κάποιες προτάσεις που θέλουν να αποδυναμώσουν το σχέδιο της οδηγίας. Γιατί Είπαμε ότι μία αποδυναμωμένη οδηγία δεν θα έχει πλέον νόημα. Ένα άλλο θέμα. Αυτή η οδηγία αφορά την καταχώρηση των επιχειρήσεων. Σύμφωνο με πολλές ε, από τις ε, παρατηρήσεις σας, όμως ε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της λειτουργίας και της εγγραφής των επιχειρήσεων. Επίση, τα έγγραφα από τον οποίο εργαζόμαστε τώρα στην Επιτροπή Γιούρη, που αφορούν το εταιρικό δίκαιο, δεν αποτελούν δεσμοί μέτρων, είναι ξεχωριστά νομοθετήματα. Εγώ δεν ε, θεωρώ ότι η δική μου έκθεση αποτελεί μέρος ενός ε, πακέτου. Η κυρία Ρέγνερ έχει δικές της ε, ξεχωριστές εκθέσεις, επομένως και εγώ το βλέπω διαφορετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. είναι το σημείο 32. Στην αρχή σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να ευχηθώ χρόνια πολλά στην κυρία Ντελβό και έτσι να δημιουργήσω ένα, μια όμορφη ατμόσφαιρα και το ίδιο έχω να πω και σε εσάς συνάδελφοι. Χρόνια πολλά. Το κοινοβούλιο είναι φτωχό και δεν μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε λουλούδια. Λοιπόν, κύριε Λεμπρετόν, εσεί που έχετε γενεθλία σα σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με ευχηθήκατε χρόνια πολλά. Ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Ωραία έκπληξη. Και εγώ εύχομαι χρόνια πολλά στην κυρία Ντελβό. Ότι καλύτερο θα σα το φοβούν έτσι καλώ γιατί το ήξερα πριν. Ε, είδατε, σα έκοψα την όρεξη γιατί προηγήθηκα, λέει ο πρόεδρο. Εντάξει, να ξέρετε όμω ότι το εννοώ. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη που εξαρτάται από την Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι σημαντικό όμως και η Νομική Επιτροπή να γνωμοδοτεί για το σχέδιο κανονισμού αυτό. Συχνά επιμένουμε στην οικονομική διάσταση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτιστική διάσταση είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο σημαντική από την οικονομική. Στην αρχή, λοιπόν, δώσαμε προτεραιότητα στην οικονομική διάσταση. Αυτό θέλαν και οι πατέρες, ο Ζαμονέ και λοιπά. Εντάξει, δεν είναι δικιά μου επιθυμία, αλλά πάση περιπτώσει. Ευτυχώ, όσο περνούσαν τα χρόνια, διαπιστώσαμε ότι δεν θα έπρεπε να γνωρούμε και την πολιτιστική διάσταση. Οπότε σήμερα έχουμε το άρθρο 3 της Συνθήκης ε, Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φροντίζει να προάγει την πολιτιστική κληρονομιά. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα σημαντικό στόχο που έχει η Ευρώπη μας. Το πρόγραμμα αυτό, Δημιουργική Ευρώπη, άρχισε το 2014. Στην πραγματικότητα συγκέντρωνε άλλα παλιότερα προγράμματα που ήδη υπήρχαν, δεν ήταν κάτι εντελώ νέο, με ένα δισεκατομμύριο 460 εκατομμύρια για την περίοδο 2014-2020. Και προβλέπονταν ε, μία αύξηση 1 δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια για την ε, περίοδο 2025. Υπάρχουν δύο υποπρογράμματα. Το ένα είναι το, πρόγραμμα, το υποπρόγραμμα Media που στηρίζει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης με διάφορες δράσεις που χρηματοδοτούνται, κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση οπτικοακουστικά, χρηματοδότηση οπτικοακουστικών ε, προγραμμάτων, ακόμα και βιντεοπαιχνίδια όχι μόνο δηλαδή με την παραδοσιακή έννοια. Διευκολύνει προγραμματισμό τηλεοπτικών προγραμμάτων, επίσης στηρίζει την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, ε, φεστιβάλ κινηματογράφου. Αυτό λοιπόν το υποπρόγραμμα Media είναι και το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Πρόκειται για το 56% του προπολογισμού. Το δεύτερο υποπρόγραμμα είναι πολιτισμικό. Ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή πολιτιστική ανάπτυξη σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται δηλαδή για την πολιτιστική συνεργασία, δημιουργία πολιτιστικών ευρωπαϊκών δικτύων, ευρωπαϊκές ε, πολιτιστικές ε, πλατφόρμες, ε, προγράμματα λογοτεχνικής μετάφρασης με 31% του συνολικού προϋπολογισμού. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται αφού προηγουμένως προσφύγουμε στις δημόσιες αγορές. Βέβαια 56 και 31 λείπει ένα 13% και αυτό το 13% είναι για τη χρηματοδότηση αυτού που ονομάζεται διατομιακός κλάδος ουσιαστικά χρηματοδοτούνται έτσι γραφεία. Και γιατί, γιατί χρειάζεται μια υπηρεσία για να προχωρήσουν τα προγράμματα αυτά που ασχολείται με τα οπτικοακουστικά και τον πολιτισμό. Και στην κάθε χώρα που συμμετέχει κανονικά υπάρχει ένα γραφείο που είναι της Δημιουργικής Ευρώπης και το οποίο έχει ως κύριο καθήκον να ενημερώνει για το πρόγραμμα, να βρίσκεται κοντά στον κόσμο δηλαδή και να τον ενημερώνει για το πρόγραμμα. Και στη συνέχεια δεύτερο καθήκον είναι να ετοιμάζει τους φακέλους των υποψηφιωτήτων. Έχει και κάποια γραφειοκρατία το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε. Μπορεί κανείς να τα βάλει με την βαριά αυτή διαδικασία, αλλά τι να κάνουμε. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, Ισλανδία, Νορβηγία, Αλβανία, Βοσνία, Μακεδονία, Ευρωμούνη, Σερβία. Η Τουρκία όμως αποσύρθηκε από το πρόγραμμα. Γενικά, το πρόγραμμα αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. έχουμε πολύ περισσότερες υποψηφιότητες πρώτα απ' όλα από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Άρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον παραπάνω από αυτό που μπορεί να καλυφθεί. Γι' αυτό και προβλέπεται αύξηση στον προπολογισμό. Και υπάρχουν και μεγάλες επιτυχίες. Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου είναι μια επιτυχία. Ή η, η ορχηστρα Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας με κάθε μετριοφροσύνη εμείς θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε κάπως τα πράγματα με τη γνωμοδότησή μας. Νομίζω ότι πρέπει εδώ να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στο πρόγραμμα και την πνευματική διοκτησία. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό ακόμα. Και γιατί, γιατί στηρίζουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό όχι μόνο με οικονομική ενίσχυση, αλλά και με νομικά εργαλεία και μέσα. Κάτι το οποίο δεν το λαμβάνει υπόψη αρκετά το πρόγραμμα. Ενώ δηλαδή την προστασία της πραγματικής ιδιοκτησίας. Άρα πρέπει να το πούμε. Ήδη αν πετύχουμε σε αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο. Δηλαδή είμαστε στην ψηφιακή εποχή και δημιουργούνται όλο και πιο μεγάλα προβλήματα για τη διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε σχέση με την ανταγωνιστικότητά μας. Και εδώ θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Το Amazon, το Netflix αρχίζουν να παράγουν τις δικές τους ταινίες και έχουν φυσικά τεράστια δύναμη. Μπορούν να κυκλοφορούν στον κόσμο ολόκληρο τις παραγωγές τους, κάτι το οποίο μπορεί να απειλήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία κινηματογράφου. Υπάρχουν κάποια νησιτικά στοιχεία για τη Γαλλία, για παράδειγμα. Το ποσοστό γαλλικών ταινιών λιγότερο από ένα στα δύο που κυκλοφορεί στη Γαλλία σήμερα ε, αποδίδει οικονομικά. Το 12%. Αν λοιπόν ήδη έχουμε κάποιες δυσκολίες και έχουμε από την άλλη μεριά τα φαινόμενα αυτά που σας περιέγραψα τα ψηφιακά από μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που γεμίζουν το κενό, καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος αυτός πρέπει να επισημανθεί στο κείμενο που ετοιμάζουμε. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε τις συμπαραγωγές. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι όταν ε, υπάρχει συμπαραγωγή από δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκές χώρες, περνάει τα σύνορα και κυκλοφορεί το προϊόν αυτό πολύ πιο εύκολα από ό,τι η παραγωγή γίνεται από μία μεμονωμένη χώρα. Έχουμε πολλά παραδείγματα συγχρηματοδότησης. Υπάρχει μια μεμονωμενη χωρα εχουμε πολλα παραδειγματα συγχρηματοδοτηση υπαρχει μια ταινια που ονομάζεται Fox Trot. Εγώ δεν την είδα, οπότε δεν λέω ότι σα τη συστήνω. Πάντω βγήκε το Μάιο του 2018 και είναι γαλλογερμανική ταινία συμπαραγωγή. 80% των ευρωπαϊκών ταινιών είναι εθνικές παραγωγές. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πολλά μπορούν να γίνουν υπέρ συμπαραγωγών και συγχρηματοδότηση ταινιών. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Τι άλλο. Μια τρίτη διευκρίνηση που θέλω να κάνω. Πρέπει να διευκρινιστούν κάποιες έννοιες που χρησιμοποιούνται. Τι σημαίνει κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης, που είναι το άρθρο 6. Τι είναι αυτό. Νομίζω ότι αυτή η έννοια θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί περισσότερο. Κυρίως όταν θέλουμε να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση. Στην αιτιολογική σκέψη αναφέρεται κάτι γι' αυτό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι σημαίνει παραπληροφόρηση ακριβώς. Ο πολιτισμός, θέλω να πω, είναι ποικιλομορφία, πολυμορφία το να θέλουμε να προωθήσουμε μια πληροφορία που θέλουμε να θεωρούμε αληθή σε βάρος μιας άλλης μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Οπότε αυτή η κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης θα ήθελα να το ψάξουμε περισσότερο τι ακριβώς σημαίνει. Και υπάρχει και μια άλλη έννοια που είναι ενδιαφέρουσα, είναι η κοινωνική ένταξη που αναφέρεται πολλές φορές στο άρθρο 4Γ για παράδειγμα. Έχει ηχθεί πολύ μελάνε στη Γαλλία από τους νομικούς, γιατί υπάρχει κάτι επίσημο που είχαμε το 2013 που μιλούσε υπέρ αυτής της έννοιας. Και ήταν μια ειλικρινή έκθεση, έδειχνε ότι η ένταξη δεν είναι το ίδιο με την αφομοίωση ε, ότι η αφομοίωση που πολλές φορές ήταν το μοντέλο της γαλλικής δημοκρατίας Σημαίνει ότι ο μετανάστης που έρχεται και γίνεται Γάλλος εξορισμού υιοθετεί πλήρω τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, τη γαλλική, το γαλλικό δηλαδή πολιτισμό και κουλτούρα και νοοτροπία, γίνεται δηλαδή πλήρως Γάλλος και μάλιστα χάνει ακόμα και τη μνήμη του πολιτισμού της χώρας προέλευσής του. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Έτσι, στην Τρίτη Γαλλική Δημοκρατία ήταν αυτό το παραδοσιακό μοντέλο. Υπάρχει ένα άλλο μοντέλο που το αντικατέστησε και που κυριαρχεί σήμερα στη Γαλλία, που είναι αυτό που λέμε ένταξη. Δηλαδή ζητάμε από αυτόν που θέλει να κατασταθεί στη Γαλλία να προσαρμοστεί στο πολιτισμό της χώρας υποδοχής, αλλά διατηρώντας σχέσεις με την χώρα προελευσής του και τον πολιτισμό της. Και υπάρχει βέβαια και εκείνο της συμπερίληψης, πώς να το πούμε, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, γιατί υποχρεώνει και τις δύο πλευρές να προβούν σε κάποιο είδους διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την οποία και η χώρα υποδοχής και ο μετανάστης βρίσκουν έναν τρόπο συνύπαρξης δεχόμενοι ο ένας τα, τον πολιτισμό και τις συνήθειες του άλλου. Δεν είναι αυτό που επιθυμώ εγώ. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι ένα πολύ επικίνδυνο μοντέλο αυτό για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οπότε πρέπει να το χτενίσουμε λιγάκι εδώ το λεξιλόγιο. Το κείμενο το οποίο έχουμε εδώ χρησιμοποιεί τον όρο inclusion. Η ιδεολογική σκέψη 11 αναφέρει και τις δύο έννοιες. Μια τη μία, μια την άλλη. Εγώ νομίζω ότι εδώ πέρα οι λέξεις έχουν τη σημασία τους και η γλώσσα δημιουργεί κάποιους συμβολισμούς και δημιουργεί πολιτική. Επίσης, κάτι άλλο, εντάξει δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά πραγματικά με εκπλήσει εδώ η σημασία που δίνεται στις κατεξουσιοδότηση πράξης της Κομισιόν. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 4. Μια που δεν είναι και πολύ μεγάλος ο κανονισμός, το κεφάλαιο 4 είναι μεγάλο παρόλα αυτά. Και έχουμε την αίσθηση ότι τελικά το σημαντικό σε αυτόν τον κανονισμό είναι κατεξουσιοδότηση πράξης. Ας επωφεληθούμε από αυτή την ευκαιρία για να σκεφτούμε λίγο τι συμβαίνει και να πλαισιώσουμε, αν μη τι άλλο, αυτό το δικαίωμα της Επιτροπής της Κατεξουσιοδότηση Πράξης. Εγώ καλλιώς πιστεύω ότι είναι κάτι υπερβολικό. Αν θέλουμε ένα δημοκρατικό μοντέλο, θα πρέπει όσο γίνεται περισσότερο να αποφύγουμε την εξουσία της γραφειοκρατίας, όπου και αν βρίσκεται αυτή, ακόμα και στην Επιτροπή. Και σας ευχαριστώ που ακούσατε τις σκέψεις μου. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεμπρωτών. Ο κύριος Ζουτόφσκι έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, Οι καλλιτέχνε και ο δημιουργικό τομέα τη Ευρώπη χρειάζεται τη στήριξή μα. Η πρόταση τη Επιτροπή επιτρέπει τη συνέχιση του προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη ε, στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο περιπολογισμό αυτή τη φορά είναι μεγαλύτερος από ότι στο προηγούμενο πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο και σίγουρα θα συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Η τεχνολογική επανάσταση επέφερε μεγάλες ε, δυσαναλογίες ε, στην Ευρώπη, ιδιαίτερα Προ όφελο του οπτικοακουστικού περιεχομένου από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Χρειάζεται οι δημιουργοί στην Ευρώπη να επιταχύνουν έτσι ώστε να μπορέσουν να συναγωνιστούν ε, την, ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε, την παραγωγή ε, τέχνης, ε, οπτικοακουστικού περιεχομένου, μουσικής κτλ. Θέλουμε να ενισχύσουμε τους ε, δημιουργούς με μικρό δυναμικό τους, δημιουργούσε μικρή κλίμακα. Η ποιότητα της ε, δουλειάς τους θα πρέπει να είναι εκείνη που θα καθορίζει ποιος θα ενισχυθεί οικονομικά και ποιος όχι, παρά οι οικονομικές προβλέψεις. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει δική μεταχείριση για κάποιες ε, περιπτώσεις χωρίς να χρειάζεται εκείνοι να ε, υποβάλουν πρόταση. Αυτό όμως δεν μας βρίσκει σύμφωνος διότι θεωρούμε πως ε, πρέπει η πρόταση να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Θα υποβάλουμε τις δικές μας τροπολογίες γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ σύντομα αν έχετε κάτι να πείτε. Όχι. Ωραία. Δεν τολμάτε. Μετά την παρουσίαση του εισηγητή ίσως αλλά τέλος πάντων εμείς ευχαριστώ να σας ακούσουμε. Κύριε Λεμπρετών, θέλετε εσεί κάτι να πείτε για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Όχι πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Απλώς ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σα για τα γενέθλιά μου. Είναι και αυτό μέρος του πολιτισμού, έτσι. Είναι καλή αγωγή. Προέδρο. Ναι. Δύο λόγια θέλω να πω κι εγώ. Το ζήτημα που εξετάζουμε είναι θεμελιώδες. Στην Ευρώπη δεν λέμε ότι η δημιουργία είναι κάτι παραπάνω από 530 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στη δημιουργία, παραπάνω από ό,τι στην αυτοκινητοβιομηχανία και ε, τη... πληροφορίες μαζί τα telecom. Οπότε γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία το θέμα, κυρίως τώρα που είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Συγγνώμη για αυτή την παρέμβαση, αλλά ήθελα να το έχω πει. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Λεμπρετών. Περνάμε στην κυρία Κάφμαν, αλλά η κυρία Κάφμαν είπε ότι δεν θα μπορέσει να είναι εδώ. Ζητά συγγνώμη. Να πούμε πότε είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών τουλάχιστον, 15 Οκτωβρίου. Έτσι, ωραία. 15 Οκτωβρίου για τις τροπολογίες. Σημειώστε το. Επόμενο σημείο ήταν το δικό μου το οποίο αναβλήθηκε. Και έτσι φτάνουμε στην ανταλλαγή απόψεων για το κείμενο της κυρίας Μπερζερόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μπερζερόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ σύντομα θα σας παρουσιάσω την θέση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί μια οδηγία της 16 Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία των ε, αυτοκινήτων και τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής. Αυτή η πρόταση οδηγίας έχει ως στόχο να απαντήσει καλύτερα στις ε, νέες απαιτήσει της ε, προστασίας των θυμάτων τροχαίων σε ένα κράτος που είναι διαφορετικό από αυτό της κατοικίας ή σε περίπτωση που έχουμε έναν οδηγό που προέρχεται από ένα κράτος μέλος η οδηγία του 2009 που έχει κωδικοποιηθεί ε, που έχει κωδικοποιήσει άλλες πιο παλιές οδηγίες έρχεται να ενισχύσει την ε, νομοθεσία και καθιστά ε, την ασφάλεια της αστικής ευθύνης για κυκλοφορία των αυτοκινήτων υποχρεωτική. Μετά το 2009 είχαμε διάφορες δυσκολίες για οι δύο τεχνικούς λόγους. Νομίζω ότι είχε μείνει ανοιχτό κάποιο μικρόφωνο ίσως του κυρίου Λεμπρετών και υπήρχε μια δυσκολία. Ε, donc, je Μάλιστα, από το 2009 εμφανίστηκαν πολλές δυσκολίες στον τομέα. Η Κομισιόν μέσω μιας εξελόγησης της εφαρμογής αυτής της οδηγίας ότι έπρεπε να προσαρμοστεί σε κάποια σημεία προκειμένου να εγγυηθεί τον κύριο της στόχο, δηλαδή την προστασία των θυμάτων, ε, των ατυχημάτων σε διασυνοριακό επίπεδο. Το κείμενο που μας παρουσιάζεται σήμερα τροποποιεί την οδηγία του 2009 σε πέντε ουσιαστικά σημεία. Το πεδίο εφαρμογή της οδηγία είναι το άρθρο 1, η οδηγία του 2009, ο έλεγχος ε, των ε, πολλαπλασιάζεται και αφορά το άρθρο 4, πάντοτε στην οδηγία του 2009, εναρμόνιση για να θεωρήσει το ελάχιστο ποσού κάλυψη, άρθρο 9 της οδηγια ε, το θέμα τη περιπτωση που είναι αφαιρέγγυο η ασφαλιστική εταιρεία, άρθρο 10, και η τροποποίηση και ε, η ανάληψη του καταλόγου των ζημιών. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η οδηγία διορθώνει την, ε, τα κενά δικαίου σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, έλεγχο της ασφαλιστικής κάλυψης ε, έπρεπε ε, να υπάρχει μια απαγόρευση των κρατών να ελέγχουν την ασφαλιστική κάλυψη για αυτοκίνητα που δραστηριοποιούνται κυρίω σε επικράτειες άλλων κρατών μελών και να μπορούν στη δική τους επικράτεια να κάνουν ελέγχους απαραίτητους και αναλογικούς που δεν θα είναι δυσδυτικοί αυτή είναι μια νέα διάταξη που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Γιατί καταπολεμάται ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα από εσά, σε περίπτωση που έχουμε υλικέ ή σωματικέ ζημίε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη νέα πρόταση, στο βαθμό που τα κράτη μπορούν να πάνε πέρα από αυτό το ελάχιστο ποσό και αυτά τα ποσά θα είναι ε, αντικείμενο πενταετού αναθεώρηση ε, βάσει ερμονισμένου δημοσίου περίπτωση αφαιρεγκαιότητα του ασφαλιστή ε, και βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε μακρές διαδικασίες αποζημίωσης. Η πρόβλεψη ενός ταχαίως μηχανισμού είναι μεγάλο βήμα προς τα μπρος. Η πρόταση έχει συμπεριλάβει την πρόταση σε κάθε κράτος μέλος ενός ταμείου αποζημίωσης ε, που ε, ουσιαστικά καλύπτει την περίπτωση που είναι αφαιρέγγιος ο ασφαλιστής σε διασυνοριακή υπόθεση. Άμεσα θα αποζημιωθεί το θύμα από το κρατικό ταμείο ε, πριν αυτό να αποζημιωθεί από το Ταμείο του Αφαιρέγγιου Ασφαλιστή. Αυτό το σύστημα υπάρχει ήδη σε πολλά και το γεγονός ότι προβλέπουμε να να υπάρξει σε όλα τα κράτη-μέλη με εκούσιο τρόπο αποτελεί σημαντική πρόοδο, γιατί από εκεί περνάει η προστασία των θυμάτων. Η ε, Κομισιόν θέλει να ενθερίνει. Συγγνώμη που σας ενοχλώ και πάλι. Υπάρχει ουσιαστικά ένας αντίλαλος, υπάρχει κάποιο μικρόφωνο ανοιχτό. Κάπου κοντά σας. Μήπως είναι τα ακουστικά σας. Τα ακουστικά σας έχουν ε, αυτή τη συνεπία. Απλώς να σας πω ε, ότι παρόλο που βιαζόμαστε, ναι, ξέρω, μιλάω πολύ γρήγορα, λέει η μιλήτρια. Λοιπόν, η Κομισιόν θέλει να ενθαρρύνει το να λαμβάνεται ε, υπόψη ή κατάλογοι των ζημιών προκειμένου να ε, υπάρχει εναρμόνιση αυτών, με βρίσκει σύμφωνη. Ο στόχος είναι να έχουμε λιγότερες απάτες και περισσότερη διαφάνεια ε, μέσω της ε, ταυτοποίησης αυτών των καταλόγων ζημιών. Ε, η πρώτη φορά το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Εγώ υποστηρίζω τη βούληση της Κομισιόν να κωδικοποιήσει την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τουλάχιστον να υπάρχει ένας ορισμός σε ό,τι αφορά την έννοια της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ περιοριστικός ο ορισμός που έχει επιλεχθεί και αποκλίνει έναν αριθμό οχημάτων, γιατί συνήθως ε, χρησιμοποιούνται ως μέσα μεταφοράς, αλλά μπορούν να προκαλούν ατυχήματα. Και παραθέτω ακριβώς αυτόν τον ορισμό δεν ε, ξέρω αν υπάρχει σε κάτι άλλε νομοθεσίες, αλλά παραδείγματο χάρη ένα όχημα που έχει κινητοποιηθεί σε μία οδό δεν είναι ένα συνηθισμένο μηχανοκίνητο όχημα ε, που κυκλοφορεί στο δρόμο και δεν μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται κυρίως στο κατασκευαστικό τομέα, στα δημόσια έργα και έχουν διασυνοριακές δραστηριότητες μπορούν επίσης να προκαλέσουν ατύχημα. Θεωρώ ότι ο ορισμό που έχει επιλεγεί ε, αυτό δηλαδή τη κυκλοφορία των αυτοκίνητων πρέπει να είναι στο δυνατόν πιο ευρύ, προκειμένου να έχουμε τόσο δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των θυμάτων ατυχημάτων. Ο στόχο εδώ είναι να προστατεύσουμε ε, τα θύματα των ατυχημάτων και να μπορούν να λάβουν αποζημίωση χωρί να έχουμε πολύπλοκε διαδικασίε και να βρούμε ποιο είναι ο πραγματικό υπεύθυνο του ατυχήματο. Έχω καταθέσει τροπολογία στο σημείο αυτό, μπορεί να τη διαβάσω αν σα ενδιαφέρει και φυσικά περιμένω να ακούσω και τα δικά σα σχόλια για το θέμα αυτό και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Merci Σας ευχαριστούμε. Συγγνώμη που σας διέκοψα δύο φορές. Ποιος θέλει το λόγο για το θέμα αυτό, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, οι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν στην Οδηγία 123 έχουν στόχο να βελτιώσουν την προστασία όσων ε, πλήττονται από τροχαία ατυχήματα και να βελτιώσει την ε, ροή της κυκλοφορίας. Ενισχύει την κοινή αγορά της οδικής ασφάλειας και αυξάνει το επίπεδο προστασίας των ε, θυμάτων επιτρέποντάς τους να λάβουν πλήρη αποζημίωση παρά το γεγονός ότι ορισμένα ε, ότι αν το ατύχημα συμβεί σε άλλο, κράτο, σε κράτος μέλος δεν δέχεται το κράτος να καταβάλει αποζημίωση. Το ελάχιστο εγκείμενο ποσό είναι ένα τομέα που θα πρέπει να εναρμονιστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει μια ελάχιστη προστασία για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Στην πρόταση όμως δεν μας ικανοποιεί ο πολύ ευρύς ορισμός της κίνησης των οχημάτων ή η επαλήθευση της περίοδου ασφάλισης, ακριβώς διότι οι ασφαλιστές εφαρμόζουν ε, διαφορετικά κριτήρια. Και σύμφωνα με αυτό χρεώνουν διαφορετικά ασφάλιστρα. Και εγγύησεις επίσης. Η πρόταση συμφωνα με αυτο χρεωνουν διαφορετικα ασφαλιστρα και εγγυησης επισης η προταση ειναι για 12 μόνο μήνες, αλλά νομίζω σαφ και ελπίζω να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν παρακαλώ θέλει το λόγο. Και ποιος ε, παρακαλώ είναι αρμόδιος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό, για το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες και για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς αλλά και υποστηρίζει το σύστημα του Σέγγεν όλας. Όπως αναφέρουμε στην ανάλυση της οδηγίας, σε, στο 99% των περιπτώσεων ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς προτείνουμε όμως αυτή τη μικρή βελτίωση έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν κάποιες πρακτικές δυσκολίες που ανακύπτουν. Αυτή είναι νομίζω η ουσία της πρότασής μας. σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα σημεία που αναφέρθηκαν από την εισηγήτρια, να πω πως δεν ακόμα συχνά ότι ο ορισμός που προτείνουμε για τον χρήστη του οχήματος είναι περιορισμένης σημασίας. Είναι ευπρόσδεκτο το σχόλιο αυτό, καθώ και οποιαδήποτε πρόταση για αύξηση τη προστασία των οδηγών. Αυτό όμω είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασιστεί σε διαπραγματεύσει, γιατί για παράδειγμα ακούμε ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογή σε ιδιωτική περιουσία, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν ανήκουν εκεί. Γι' αυτό λοιπόν ε, νομίζω πω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι ανταλλαγέ απόψεων και πρέπει να ακούσουμε όλε τι απόψει. Μετά αναφέρθηκε το ελάχιστο ποσό κάλυψης. Καθώς και ένα πρόβλημα με τα πιστοποιητικά και το ιστορικό των αξιώσεων. Εμείς θέλουμε να επιτύχουμε το ελάχιστο δυνατό επίπεδο προστασίας χωρίς να παρεμβαίνουμε στα κριτήρια κινδύνου που έτουν οι ασφαλιστικές εταιρείε. Αυτό το βασίζουμε στην ε, ρήτρα απαγόρευση των διακρίσεων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα θέταμε σε κίνδυνο τα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών εταιριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις απόψεις σας τις προτάσεις σας. Ελπίζω οι διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν γρήγορα έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε έξισου γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Η κυρία Μπερζερόν τότε για να ολοκληρώσουμε το θέμα, αν έχει κάτι να προσθέσει. Όχι, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Πράγματι, πρόκειται για ένα καλό κείμενο το οποίο βελτιώνει την προστασία των χρηστών και των θυμάτων ατυχημάτων. Είναι ένα πολύ καλό κείμενο το οποίο εναρμονίζει την νομοθεσία. Όντω πρέπει να συμφωνήσουμε για του όρου, την ορολογία. Είναι θέμα σημαντική και είναι και το θέμα τη Ευρώπη αυτό. Πρόεδρος, ναι, ένα τεράστιο θέμα που δεν θα κλείσει σίγουρα σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ. Επόμενο θέμα είναι το σημείο 36 που ήταν ανταλλαγή απόψεων ε, με τον κύριο Σβόποντα, ο οποίο όμω δεν μπορεί να είναι εδώ, έχει αναβληθεί αυτό το σημείο. Σημείο 37 στην ημερήσια διάταξη είναι η παρουσίαση του κύριου Κοφεράτη. Η κυρία Γκούντελαντ θα μας το παρουσιάσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Γκούντελαντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Κοφεράτη, τα συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι εδώ, έπρεπε να φύγει από τι Βρυξέλλες νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει λόγω κάποιων ανελημμένων υποχρεώσεων στην πατρίδα του. Θα διαβάσω επομένως τις απόψεις του κυρίου Κοφεράτη. Ο κύριος Κοφεράτη θα ήθελε να ευχαριστήσει τους κοιόδης εισηγητέ και τους συναδέλφους προκαταβολικά για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην πρόταση κανονισμού για την επίδοση δικαστικών εγγράφων. Θα δεχτεί όλες τις προτάσεις και τα σχόλια για το σχέδιο έκθεσης. Όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός για την επίδοση δικαστικών και εξώδικων εγγράφων σε αστικές εμπορικές υποθέσεις είναι ουσιαστική σημασία για την διασυνοριακή δικαστική συνεργασία και για θέματα του αστικού εμπορικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια πρόταση να τροποποιηθεί ο κανονισμός ε, και να γίνει σε βάθος αξιολόγηση με στόχο πιθανές βελτιώσεις. Ο κύριο Κονφεράτη στηρίζει το στόχο της Επιτροπής να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των ε, δικαστικών δικαστικών σε ό,τι αφορά την επίδοση δικαστικών και εξωδικών εγγράφων. Θεωρεί πως ε, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των ε, διαδίκων και πως η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα έχει υψηλά πρότυπα ασφαλεία και προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Κοφεράτη ζητά, ένα, ζητά το σύστημα πληροφορικής που θα χρησιμοποιηθεί να βασίζεται στον ε, e-codex και οι λεπτομέρειες που θα τον διέπουν να καθοριστούν με καταξιοδότηση πράξης. Επίσης, ε, είναι υπέρ της ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφων, όμως για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του εναγόμενου, είναι πολύ σημαντικό να ε, υπάρχει ρύθμιση των υπηρεσιών. Επίσης, η επίδοση εγγράφων σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ε, θα πρέπει να συνοδεύεται και από το δικαίωμα του να να ορίζει κάποιον εκπρόσωπο που θα λαμβάνει τα έγγραφα αυτά, όμως αυτό δεν ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ιδιαίτερα για να αποφύγουν πρόσθετο κόστος. Ο κύριος Κοφεράτη θεωρεί επίσης ότι το κόστος των ετούντων για πρόσβαση σε δικαστικές οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να είναι προβολικό και αυτό για τρεις λόγους. Είναι απαραίτητο καταρχάς να Υπάρχει όριο, στις, ε, ανά όριο στις, ε, στο κόστος που επιβάλλουν τα κράτη-μέλη και στα τέλη έπειτα για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο. Τέλος, το σχέδιο έκθεσης. Ο εισηγητής προτείνει την εισαγωγή ορισμένων διευκρινήσεων και μικρών αλλαγών, μεταξύ άλλων τις ε, προθεσμίες για ε, μεταδόση, διαβίβαση πληροφοριών στις ε, διάφορες υπηρεσίες. Δεύτερον, την δυνατότητα του εκείνου που λαμβάνει το έγγραφο να αρνηθεί να το λάβει σε περίπτωση που είναι σε γραμμένο σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνει και έπειτα να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εναγόμενων σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ο κ. Κοφεράτη σίγουρο ότι η συνεργασία με τους Κιώδη και τους υπόλοιπου συναδέλφου θα είναι πάρα πολύ καλή και, για... και με το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Ο κ. Κοφεράτη θα χαρεί πολύ να λάβει τα σχόλια και τις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ. Έχει... Είναι πολύ τυχερός που εσείς τον εκπροσωπήσατε εδώ. Λοιπόν, θέλει κανεί το λόγο. Όχι, δεν βλέπω κανέναν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε, εφόσον επιθυμεί. Έχει σχόλια. Όχι. Όχι. Όχι σχόλια. Όχι κομισιόν. Ωραία. Ε, κύριε Γκούντελαντ, κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι. Καλώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το θέμα. Α, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, ναι. 24 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Εντάξει. Επόμενο σημείο. Ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Ράντεφ, ο οποίος όμως έπρεπε να φύγει το πρωί γρήγορα. Οπότε θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από κάποιο άλλο συνάδελφο που δεν είναι μέρος τη Ιουρή να παρουσιάσει την έκθεσή του, αλλά είναι οριακό. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να αναβληθεί. Παρακαλώ όμως. Εσείς. Και πάλι ο κύριος Κοφεράτη θέλει να πει δύο λόγια για αυτό το θέμα και θα μιλήσω εκ μέρους του αν συμφωνείτε. Α, αναβλήθηκε. Α, εντάξει τότε. Καλώς. Κοιτάξτε, κύριε Γκούτελαντ, θέλαμε να διευκρινίσουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που είναι 24 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η κυρία 22, λέει κύριε Γκούτελαντ. Α, 24, 24 λέτε. Καλώς. 24 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Το εξαντλήσαμε, αναβάλαμε το σημείο του κυρίου Ράντεφ. Οπότε φτάνουμε τώρα στο σημείο 39 που μας παρουσιάζει ο συνάδελφος κύριος Χρυσόγονος. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Merci, merci, le président. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επιτυχία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία και κατά πόσο θα διασφαλίσει υψηλά επίπεδα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, κοινωνικής συνοχής, χωρίς αποκλεισμούς, με δραστηριοποίηση στην κοινωνία. Για να υπάρχει αυτή η ανταγωνιστικότητα, η αντοχή της Ευρώπης και η συνοχή στην Ευρώπη σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους, στην υγεία τους, στην εκπαίδευση και στην δημιουργία. Παρά τις κάποιες βελτιώσεις, η μακροχρόνια ανεργία, όπως και η ανεργία των νέων, βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη. Αυτοί που κινδυνεύουν από φτώχεια στην Ευρώπη, από κοινωνικό αποκλεισμό, είναι πάρα πολλοί. Επιπλέον, υπάρχουν οι δημογραφικές τάσεις, η γύρανση δηλαδή του πληθυσμού ή οι μεταναστευτικές ροές που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί ένα κατεξοχή οικονομικό εργαλείο για να βελτιώσει την κινητικότητα των εργαζομένων και τις ευκαιρίες απασχόλησης, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή, τη δικαιοσύνη, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και μειώνει ανισότητες, άδικες και άχρηστες μεταξύ των χωρών μελών. Με επιπλέον προϋπολογισμό 101 εκατομμυρίων ευρώ για 7 χρόνια, 2021 με 2027, το ταμείο αυτό συγχωνεύει το τωρινό κοινωνικό, την πρωτοβουλία για την νεολαία, το Ταμείο για την Βοήθεια για τους Πιο Φτωχούς, το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Υγεία η πρόταση συγχώνευσης όλων αυτών των ταμείων σε ένα μόνο εργαλείο υπόσχεται να λειτουργήσει ως μόχλευση για να υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος στον κόσμο, να βοηθήσει περισσότερο και να βελτιώσει και τα αποτελέσματα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Είναι, πιστεύω, ενθαρρυντικό που υπογραμμίζει τις ίσες ευκαιρίες για όλους, που αντιμετωπίζει το θέμα των ανισοτήτων στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και στην υγεία. Άλλες αλλαγές τώρα όσον αφορά το ταμείο αυτό. Μεγαλύτερη ευθυγράμμιση και συμμόρφωση προς τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και βάσει των αρχών του κοινωνικού πυλώνα για κοινωνικά δικαιώματα. Ε, ευρύτερο πεδίο εφαρμογή με αναφορές σε ηλική βοήθεια προς τους μετανάστες και μέτρα κοινωνικής ένταξης. Μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση, γιατί περιλαμβάνεται και το Ταμείο Βοήθειας προς τους πιο φτωχούς. Απλοποιούνται υποχρεώσεις των χωρών μελών ελέγχου και μειώνεται ο αριθμός των δικτών. Έτσι διευκολύνεται ο συνδυασμός των διατάξεων για την ηλική και άλλη βοήθεια για να στηριχθεί η κοινωνική ένταξη με συγκεκριμένα μέτρα. Θα υπάρχει έτσι και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις θεματικές απαιτήσει για να προσαρμοστούν στις ανάγκες των χωρών. Έτσι, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν κανονισμό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Βέβαια, παρά τις θετικές τάσεις πρέπει να γίνουν περισσότερα για να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη, η μείωση της φτώχειας και των διακρίσεων, αλλά και η προώθηση της απασχόλησης κατά από καλές Η προτερότητα δράσεων πρέπει να καθορίζεται πιο συγκεκριμένα, κυρίως σε σχέση με τον κοινωνικό πυλώνα και πάνω απ' όλα ο προπολογισμό για τέτοιε πρωτοβουλίες θα πρέπει να αυξηθεί αποφασιστικά εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πράγματα αποτελεσματικά να στηρίξει την κοινωνική ένταξη, να μειώσει τη φτώχεια και να βελτιώσει του δείχτε απασχόλησης αλλά και την εκπαίδευση. Χρειάζονται περισσότεροι πόροι προ τι χώρε μέλη που αποτελούν και τον πιο το κρίκο μερικές φορές, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία κλπ. Πρόκειται για προϋπόθεση για να υπάρχει μια Ευρώπη με περισσότερη συνοχή και βάσει αυτό το στοιχείο θα ετοιμάσω και εγώ την γνωμοδότησή μου, λαμβάνοντα υπόψη όσο γίνεται περισσότερο τις δικές σας συστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρυσόγονη. Κύριε Ντελβό έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Ρέγκνερ, που δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα στη συνεδρίαση, γιατί έχει υποχρεώσει στην Αυστρία. Θα διαβάσω, λοιπόν, τη δήλωσή της. Καταρχήν, η Αβελίν λέει ότι χρειαζόμαστε επαρκή κονδύλια για μια κοινωνική Ευρώπη. Όπως ξέρουμε, το πεδίο εφαρμογή τη σύσταση ενό ε, νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ διευρύνεται σημαντικά, η απλούστευση είναι κάτι καλό, αλλά αυτό de facto οδηγεί σε μείωση τη χρηματοδότηση τουλάχιστον κατά 10%, κάτι που είναι εντελώ απαράδεκτο για την ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών. Έτσι λοιπόν ζητάμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση, να καταπολεμήσουμε την ανέργεια, ιδίω την ανεργία των νέων, να καταπολεμήσουμε την ανέχεια, να υποστηρίξουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κυρίως όπως είπαμε σήμερα το πρωί για τις ψηφιακές δεξιότητες. Θέλουμε μέσα για τη μείωση της ανέχειας των παιδιών. Αυτό μπορεί να γίνει αν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση με ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά και δεν θα δεκτούμε μείωση στα κονδύλια για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και ε, η συγκήτρια των σοσιαλιστών ε, είναι εντελώς αντίθετη στο να συσχετιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ με τις ειδικέ συστάσεις σαν χώρα, γιατί αυτό θα οδηγήσει σε αρνητικέ συνέπειε για τους πολίτες και τους εργαζομένους. Επίσης, ε, ζητάει η κυρία Νέγκρα μεγαλύτερη έμφαση στην ισότητα ε, και στο θέμα της ισότητας των φύλων. Θα πρέπει το θέμα αυτό της ισότητας των φύλων να ενταχθεί περισσότερο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σας ευχαριστούμε που μας αναφέρετε τις απόψεις της κυρίας Ρέγνερ. Θέλετε, κύριε Χρυσόγνα, ξανά το λόγο για να ολοκληρώσετε. Σας ευχαριστώ. Είμαι πρόθυμος να ακούσω τις προτάσεις και τις τροπολογίες των υπόλοιπων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. προκειμένου να έχουν στην εδώ μεγαλύτερη ομοφωνία στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι για τις 25 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι, 25 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια ανακοίνωση ακόμη έχω να κάνω και θα, θα την κάνει η Εύα από τη Γραμματεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τις επόμενες συνεδριάσεις ε, της Επιτροπής μας θα έχουμε την ε, κοινή συνεδρίαση Λίμπε και Γιούρι στις 18 Οκτωβρίου από τις 9 στις 9.30 για την πρόταση κανονισμού που θα σπίσει το πρόγραμμα δικαιοσύνη, Justice. Υπάρχει έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο στην δεύτερη λομέλεια του Οκτωβρίου. Θα διευκρινίσουμε την ημερομηνία τις επόμενες μέρες. Και έχουμε και την τακτική συνεδρίαση στις 19 Νοεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και 20 Νοεμβρίου ολόκληρη την ημέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι όλα σαφή. Ελπίζω να μην μπερδευτήκατε με τι ημερομηνίε και τα ωράρια. Σα ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τι εργασίε μα. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα και για του δύο δυστυχεί που άλλαξαν ηλικία. Χρόνια πολλά.